Η Πρόεδρος. Ξέρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης με τα έγγραφα που έχουν εγκριθεί είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχουν παρατηρήσεις, όχι. Εγκρίνονται. Ο Πρόεδρος έλαβε την